We should start immediately because it's just half past nine or even more. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Κυρία Ντέλη, τι έχετε να μας πείτε. Καλησπέρα. Allez, s'il n'y a pas d'objection à l'ordre du jour. Αν δεν έχετε αντίρρηση με την ημερήσια διάταξη, Εγκρίνεται η μερίσια διάταξη. Να επενθυμίσω ότι είμαστε στο διαδίκτυο, εκπέμπουμε. Και κανονικά έχουμε διερμηνία σε όλες τις γλώσσες. Έχετε τη γλώσσα σας όλοι. Σχόλια υπάρχουν. Κύριε Κέλλη, τι τρέχει. Έχετε πρόβλημα. Όχι. Ωραία. Εάν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, θα ξεκινήσω μέσω στις ψηφοφορίες. Θα δώσω στον κύριο Μπούζεκ την τιμή να οργανώσει την πρώτη ψηφοφορία. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ξεκινάμε ψηφοφορία. Η τελευταία ψηφοφορία πιθανότατα με κοινή συνεδρίαση αυτής της Επιτροπής αυτή τη θητεία και δύο επιτροπές από κοινού. Το Connecting Europe Facility, το μέσο για τη διασύνδεση της Ευρώπης, οι Μαρία, Μάριανα Μαρινέσκου, Βυρκόναν και Τελίτσκα. Έχουμε μερική συμφωνία όσον αφορά το θέμα. Καλωσορίζω όλα τα μέλη των δύο κοινοβουλευτικών επιτροπών. Κυρίως καλωσορίζω την κυρία Νταλή. Θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά η ψηφοφορία σύμφωνα με ξεχωριστό ε, κατάλογο ψηφοφοριών, μία ψηφοφορία. Δοκιμαστική ψηφοφορία. Ενδεικτική ψηφοφορία, αν ξεκινήσουμε λοιπόν. Please vote, dear Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Ωραία. Νομίζω ότι λειτουργεί το σύστημα. Δεν είμαστε και πάρα πολλοί, αλλά και οι δύο επιτροπές θα έπρεπε να είναι πάνω από 100 μέλη, τέλος πάντων θα καταφέρουμε, διότι ε, έχουμε απαρτία, έχουμε την πλειοψηφία των μελών. Διαβάσω τον τίτλο. Πρόταση κανονισμού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που δημιουργεί το μέσο για τη σύνθεση της Ευρώπης, Connecting Europe Facility, οι Μάριον Ζάνκ Βαρονέσκου, Χάραν Βιρκούνεν και Πάβελ Τελίτσκα. Ψηφίζουμε στη μερική συμφωνία που, ε, στην οποία καταλήξαμε στους άτυπους μερική διαλόγους. Έναρξη ψηφοφορίας, ονομαστική ψηφοφορία βέβαια. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. περιμένουμε. Ειδική χειρονομία για σας. Περιμένουμε λοιπόν. Πέρας. Με πολύ μεγάλη πλειοψηφία όπως βλέπετε. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια σε όλους σας που επεξεργαστήκατε την εν πρόταση. Ευχαριστώ κύριε Σιγητά. Ευχαριστώ τους Σκιώδης και των δύο επιτροπών. Η κυρία Ντελή έχει το λόγο. Δίκιο έχετε που χειροκροτείτε τον κύριο Μαρινέσκου. Μπράβο. ο Σπαβερ Τελίτσκα και εσείς συγχαρητήρια. Μπράβο κυρία Βερκούνεν, και εσείς. Μπράβο, συγχαρητήρια. Να σας πω... Ε, μιλάω. Κύριε Κουράμπατσεφ, σας παρακαλώ. Λίγο σεβασμό όταν μιλάει η Πρόεδρος. Πες το. Συγχαίρω λοιπόν όλες τις ομάδες, τη διαπραγματευτική ομάδα πάνω απ' όλα. Σας χαιρετίζω που πετύχατε το συμβιβασμό του Συμβούλιο Αργά τη νύχτα επετεύχθη, αλλά ο κύριος Μαρινέσκου... Ήτανε πρωί, καλά το λέτε, ήτανε πρωί. Ιδού λοιπόν έγινε σημαντική πρόοδος. Και τι δείχνει αυτό. Ότι τα αποτελέσματα μεταξύ Επιτροπής Ήτρε και της Επιτροπής Μεταφορών είναι καρπός πολύ καλής συνεργασίας. Ευχαριστώ όλους. Έτσι, δε περαιτέρω ότι ο μηχανισμός διασύνδεσης, το Connecting Europe Facility, είναι βασικό χαρτοφυλάκιο για τα διευρωπαϊκά δίκτυα του μέλλοντος. Αλλά κυρίως ίγκη και η ώρα πλέον για την προετοιμασία προόδου στις μεταφορές. Και στην ενέργεια και στον ψηφιακό τομέα. Πρόοδος, διότι όλοι σε αυτή την αίθουσα έχουμε επίγνωση των προκλήσεων που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Συνάδελφοι, η Επιτροπή Ήτρ και Μεταφορών είναι έτοιμες για το πρώτο αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων για την Ολομέλεια η ψηφοφορία θα λάβει χώρα στην Ολομέλεια τον Απρίλιο, δεύτερη σύνοδο του Απριλίου, θα είναι η τελευταία μας Ολομέλεια, πάση περιπτώσει ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας και αν δεν έχετε άλλα θέματα Μπορούμε να διακόψουμε τη συνεδρίαση, πέρα σα και ευχαριστώ. Κύριε Μαρινέσκου, να πείτε κάτι. Α, έχω μια ερώτηση, λέει ο κ. Μαρινέσκου. Ποιος ψήφισε κατά? Κύριε Μαρινέσκου, σε αυτό το κοινοβούλιο υπάρχει ο σεβασμός της δημοκρατία όπως αποκαλείται. Μην καταγγέλλετε, μην καταγγέλλετε, μην δείχνετε τους συναδέλφους. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πέρα σας. Ευχαριστώ, αγαπητοί φίλοι. Δύο ειδήσει έχω να σας ανακοινώσω. Το πρώτο που έχω να σας πω. Κακά μαντάτα για την Επιτροπή Μεταφορών. Δεν έχω τίποτα να σας προσφέρω άλλο. Και καλά για την Ήτρε. Θα έχουμε άλλη μια ψηφοφορία μπροστά μας. Μικρή διακοπή, διάλειμμα, διαλυματάκι και θα ψηφίσουμε τα επόμενα σημεία που έχουμε στο τραπέζι. Θα ξεκινήσουμε στις 9 ακριβώς. 9. Πρώτα απ' όλα, οι συνάδελφοι της Επιτροπής Μεταφορών ας έχουν τη δυνατότητα να φύγουν, αγαπητοί μου φίλοι. Μην είσαστε και τόσο νευρικοί. Θα παρακαλούσα τους συναδέλφους της δύο επιτροπές ότι μπορούμε να ψηφίσουμε. Αυτά είναι καλά μαντάτα, αυτά είναι άριστα.